εγκρίνουμε τους ορισμούς των ε, Προέδρων των Επιτροπών και Αντιπροσωπιών. Βρίσκονται οι ορισμοί αυτοί στα πρακτικά. Αν μέχρι τώρα συνεδρίασης δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, θεωρώ πως έχουμε εγκρίνει αυτούς τους ορισμούς. Σύμφωνα με το άρθρο 74, υπέγραψα με τον πρόεδρο του Συμβουλίου 8 νομοθετικές πράξεις οι οποίες εγκρίθηκαν με την κανονική νομοθετική διαδικασία οι τίτλοι των οποίων θα δημοσιευτούν στα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης. Περνάμε τώρα στις εργασίες μας.